στο λόγο χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση της πολιτικής για να είμαστε πιο συνεπείς ε, και να είναι και πιο συνεπείς η υποστήριξή μας προς τις ε, δημοκρατικές δυνάμεις αυτών των κρατών. Πολύ ωραία. Και τώρα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο... Όχι στον κύριο Σόκολ από το ΕΛΚ, λάθος, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Ο κύριος Χαλίτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, το ε, πρόγραμμα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στέφτηκε από επιτυχία τα προβλήματα ε, των κυβερνήσεων και οι δίθεν ε, μεταρρυθμίσεις, οι ιονοί μεταρρυθμίσεις, αυτό δεν μπορεί να το θεωρούμε πρόοδο υπάρχουν πραγματικές φιλοδοξίες των πολιτών, της ε, κοινωνίας των πολιτών. Εγώ έρχομαι από μια οικογένεια που διχάστηκε από τον πόλεμο η μισή της οικογένειάς μου είναι πολίτες αυτών των κρατών και μόλις πριν από λίγο καιρό κατέστηκε αυτούς δυνατούν να έρχονται να μας επισκέπτονται χωρίς βίζα. Η επόμενη δεκαετία όμως ε, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εντατικοποίηση των θέσεών μας γιατί μιλάμε για δύο προσωπικές σχέσεις, για σχέσεις ανάμεσα στις ΜΚΟ, για ανταλλαγέ εράσμους. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίε που μπορούν να αλλάξουν αυτές τις κοινωνίες και δεν πρέπει πρέπει να στρωθοκαμιλίζουμε μπροστά σε αυτά που πρέπει να επικριθούν. Αλλά έχουμε να κάνουμε εδώ με τρεις χώρες οι οποίες ε, είναι καθοριστικές ε, για την ανατολική εταιρική σχέση, άρα χρειαζόμαστε εξυγχρονισμό της εταιρικής σχέσης. Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία αξίζουν περισσότερα, αξίζουν ε, να τους δώσουμε μία ευκαιρία. Να μην ξεχνάμε αυτές τις χώρες. Οι χώρες αυτές υπολογίζουν σε εμά και παρότι εντάξει υπήρξαν κάποιες οπισθοδρομήσεις, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τις χώρες αυτές. Σα ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τώρα έχουν το λόγο. Η κυρία Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Υπατή Εκπρόσωπη, να σε ευχαριστήσω για την συνεργασία μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Και θέλω να πω ότι θέλω να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για το μέλλον σας, για τις μελλοντικέ προσπάθειες. Έχουμε αυξανόμενο αριθμό ανησυχιών στη γειτονιά μας Νομίζω τα μηνύματα που έρχονται από το Κίσινάου είναι ανησυχητικά. Βλέπουμε οπισθοχώρηση από τις μεταρρυθμίσεις, από τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Κάποιος θα έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε αφελής βοηθώντας την επίτευξη συμφωνίας που οδήγησε σε καταδικασμένο συνασπισμό με τον πρόεδρο που άρπαξε την εξουσία. Και στη Γεωργία ο κόσμος ζητά ένα πιο δημοκρατικό και δίκαιο εκλογικό σύστημα και αντιμετωπίζουν την αστυνομία, τις αστυνομικέ δυνάμει καταστολή που χρησιμοποιούν δακρυγόνα και πλαστικέ σφαίρες. Στο Βακού, ο ηγέτη αντιπολίτευση, σε διαδήλωση, σε μία ομιλία, συνελήφθηκε, βασανίστηκε, όπω είπε, στα χέρια τη αστυνομία. Αυτό που συμβαίνει στι χώρε αυτέ είναι αυταρχικοί που προσπαθούν να, να αρπάξουν έφταστες δημοκρατίε στα χέρια του. Κάτι που διαδίδεται και σε πολιτική η ήπια στην περιοχή δεν δίνει τα ευκταία αποτελέσματα. Τι συμβουλή θα δίνατε στο διάδοχό σας σχετικά με το πώς πρέπει να εξετάσουν τη διαμόρφωση νέας στρατηγικής. Ευχαριστώ. Κύριος Μπασέσκου. Από Θα ήθελα να θέσει μια ερώτηση ο κύριος Μπασέσκου. Έχει σηκώσει μπλε κάρτα. Δέχεστε την ερώτηση του κυρίου Μπασέσκου. Κυρία Γκίλ. Μη φύγετε. Ο, δεν δέχεται. Και φεύγει. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκέτα εν ονόματι του Ρινιού. Έχετε το λόγο. Τα μικρόφωνο σας παρακαλώ. Δουλεύει. Δουλεύει ήταν ένα καθήκον και μία αναγκαιότητα. Η Ένωση, η Ένωση πρέπει να ανοιχθεί στι χώρε τη Κεντρική Ευρώπη, έπρεπε να προσφέρει και μία εταιρική σχέση στι ανατολικέ χώρε, όπου η διεύρυνση τη έκανε νέου γείτονε. Αυτή η εταιρική σχέση έχει αδυναμίε και επιτυχίε. Αλλά δέκα χρόνια μετά κάτι προφανέ βλέπουμε. Στη δική μα ανατολική εταιρική σχέση λησμονήσαμε τη Ρωσία ή πιο ακριβώ δεν θελήσαμε να τη δούμε ε, όσον αφορά, διότι τα προβλήματα που έθετε θεωρήσαμε ότι είναι ανεπίλητα. Θα πρέπει να διορθώσουμε ε, την κατάσταση διερευνώντας ε, τη δυνατότητα νέας συμφωνίας του Ελσίνκη ασφαλείας και συνεργασίας με τη Μόσχα. Θα είναι δύσκολο, θα έλεγα όχι, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και εντελώς αβέβαιο. Πρέπει όμως να αποπειραθούμε να το κάνουμε διότι στη Ρωσική Ομοσπονδία έχουμε το άλλο ημίση της Υπήρου, είναι η χώρα η πιο εκτεταμένη στον κόσμο, που είναι φτωχή και κατεστραμμένη, αλλά η δυνατότητα να ενοχλεί παραμένει πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Τόμασιτς από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τα ε, μέλη. Ε, ε, πόσο σημαντική είναι και πόσο δυναμικό υπάρχει. Αυτό έγινε σαφές στη διάρκεια της κρίσης του μεταναστευτικού. Καλύτερες σχέσεις με τους γείτονες και ισχυρότερες πολιτικές και εμπορικές σχέσεις εγγυώνται μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτού του είδους τις καταστάσεις. Στην Ανατολή υπάρχουν χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτύξει καλές σχέσεις στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρική σχέση. Ε, πάντως πόρο απέχουμε από το ενσταθερότητα, γιατί ορισμένες βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση και κάποιες διανύουν μια οδυνηρή μεταβατική περίοδο. Επίσης, εν ώψη της θέσης μας απέναντι στην Ρωσία, το ευρωπαϊκό συμφέρον ε, λέει για ανάπτυξη πλήρως ε, ε, ε, λειτουργικών δημοκρατιών, ε, κράτων δικαίου. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Τόμασιτς. Ο κύριος Σόκο θέλει να ε, σας υποβάλει ερώτηση. Τη δέχεστε? Μάλιστα. Κύριε Σόκο, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ε, ε, κυρία Τόμασιτς, είμαι πολύ ευτυχής που επενείτε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, που υποστηρίζουμε κοινά συμφέροντα και λύσεις. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ώστε να ενισχυθούν και οι πολιτικές προς τις χώρες που αναφέρατε. Μάλιστα, βεβαίως ε, πιστεύω πως πρέπει να ενισχύσουμε την θέση μας αλλά σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες που πρέπει να λάβουν αυτές τις αποφάσεις αλλά όλα τα κράτη-μέλη από κοινού. Και εγώ σας ευχαριστώ, η κυρία Πασέσκου. Ο κύριος, συγγνώμη. Ο κύριος Πασέσκου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που χτυπήθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία και έχασε την Κρυμαία και ε, εντωμεταξύ σοβεί ε, φίλος πόλεμος στην Ανατολική πλευρά της επικράτειάς της. Η πρόσβαση στη, δε στην Μαύρη Θάλασσα έχει μπλοκαριστεί. Και γιατί αυτό, γιατί η Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορεί να δεχτεί τον προσανατολισμό της χώρας αυτής που είναι ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μείνει ακέραιη η Ουκρανία θα πρέπει να αντιστηρίξουμε. θα πρέπει να βοηθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εφαρμόζαμε το σχέδιο Σταν Μάγερ θα ήταν αυτό σφάλμα γιατί θα κινδυνεύαμε να χάσουμε ε, την κυριότητα της Ουκρανίας γιατί θα γίνει ένα δημοψήφισμα μετά από την Ομοσπονδιοποίηση και στη συνέχεια μία δήλωση ανεξαρτησίας όπως στην Οσιατία, ε, στην Αυχασία και στην ε, Κρυμαία. Αυτή είναι η, τεχνική, η ρωσική τεχνική. Ε, στην Μολδαβία ισχύει αυτό το παράδοξο ότι η αντιπολίτευση αποτελείται από δύο κόμματα ε, φιλοευρωπαϊκά τα οποία όμως ε, παρατηρούν ε, την εγκαθίδρυση μιας σκληρής αυταρχικής κυβέρνησης υπό την αιγύδα του κυρίου Ντόντον. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποτελούν την πλειοψηφία να κάνουν το καθήκον του στη δημοκρατία της Μολδαβίας αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση της χώρας και προσανατολίζοντας τη χώρα προς τη Δύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Βίτανοφ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπο. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους ανατολικούς εταίρους μας ε, είναι πολιτική πρώτης προτεραιότητας, αλλά παράλληλα ε, είναι και μια πολιτική ε, που είναι παραμελημένη αυτό αφορά κυρίως τις σχέσεις των κρατών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μοιάζει να μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι φυσικοί πόροι, και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι χώρες αυτές στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι τόσο το γεωπολιτικό στοιχείο. Παράλληλα, αυτή η περιοχή είναι ε, πεδίο αντιπαραθέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Όλα αυτά τα χρόνια δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Να αναθεωρήσουμε το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, να έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα και δεύτερον, μεγαλύτερη στράτευση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θέσουμε προτεραιότητες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ε, κινδυνεύουμε να στείλουμε τις χώρες αυτές ε, στην αγκαλιά κάποιων άλλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Στρουγκάριου, παρακαλώ, για το Renew. Η απόσυρση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης στο Κινσινάου ε, σήμαινε ότι δεν ήθελε να παίξουν το παιχνίδι του κυρίου Ντοντών. Δεν ήθελαν να επάγουν ε, την δικαιοσύνη στην κυβέρνηση και στόχος επίσης ε, ήταν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ότι υπάρχει οπισθοχώρηση όσον αφορά την προσέγγιση της Ευρώπης. Οι πολίτες ε, απομακρύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν πολύ αυστηροί για την χορήγηση της μακροοικονομικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες αυτών των κρατών γιατί είναι σημαντικές οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς σημαίνει μεταρρύθμιση. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, ε, κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση και να στραφεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινάμε κάθε φορά από το μηδέν. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η πόρτα. Χρειαζόμαστε πραγματικές μεταρρυθμίσεις να στηρίξουμε για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και για το κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσανέσκι εκ μέρους του ECR. Κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμη κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, η ανατολική εταιρική σχέση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο Ίσως ε, παλαιότερα να, ε, να αποθέσαμε μεγαλύτερες ελπίδες σε αυτό το εργαλείο από ό,τι τελικά επαληθεύτηκαν. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτό το εργαλείο αποτελεί γέφυρα προς Ανατολάς και αυτές τις έξι χώρες μπορούμε τώρα να τις εντάξουμε σε, σε τρεις ομάδες. Πρώτον τους καλούς μαθητές, όπως είπε ο κύριο Χαλίσκη, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία. Μετά έχουμε ε, δύο χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία, Αρμενία και Λευκορωσία και τέλος έχουμε το Αζερβαϊτζάν που είναι μόνο του, δεν εντάσσεται σε καμία από τις ε, δύο πριν κατηγορίες. Την ε, Λευκορωσία και την Αρμενία δεν πρέπει να τις ε, αγνοήσουμε. Δεν πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη, γιατί αν το κάνουμε, τότε αυτές οι χώρες θα πέσουν στην αγκαλιά της Ρωσίας. Όταν μία χώρα ε, δείχνει ότι είναι ουδέτερη, αυτό να το εκτιμούμε. Και ε, κάνω έκκληση, απευθύνω έκκληση ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σόφκοφ. Κύριε Σόφκοφ, ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο και είπα τη εκπρόσωπο. Την ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που έκανε. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε για την πρόθεση της ανατολικής γειτονικής σχέσης είναι τόσο ισχυρό εργαλείο για τη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μαζί με όλους μας που εργαζόμαστε σκληρά ούτω ώστε οι πολίτες αυτών των χωρών να κατανοήσουν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες είναι οι μόνες αξίες που θα μεταμορφώσουν τις κοινωνίες τους και θα βελτιώσουν τις κοινωνίες τους. Θα συνεχίσουμε να το προωθούμε αυτό. Υποστηρίζω ένθερμα την ιδέα του συναδέλφου Κομπίλιους Πρέπει να εστιαστούμε επί τριών χωρών που ακόμα τρέφουν εκεί ελπίδες, ελπίζουμε να τις βάλουμε στο σωστό δρόμο. Τους έχουμε δώσει δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις, ό,τι ευκαιρίες για τους νέους τους δώσαμε. Τους δώσαμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για να δουν πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνιών τους. Ελπίζουμε ότι αυτό το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο και θα έχετε, αν συνεχίσετε αυτό το δρόμο, τους ισχυρότερους συμμάχους εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ε, συνάδελφε Μίλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μίλλερ. Κυρία Μογκερίνη, η εμπειρία που απορρέει από τη δεκαετία της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης δικαιολογεί την ανάγκη συνέχισης πολιτικής. Έχουμε τον Υπουργό Σικόσκι, τον δημιουργό αυτή τη ιδέα, Αλλά χρειαζόμαστε αποφάσει που θα ανταποκρίνονται στα νέα διλήμματα και τι νέε προκλήσει. Το βασικό θέμα είναι το μοντέλο των εταιρικών σχέσεων που οδηγούν σε μια οικονομική ολοκλήρωση και σε μικρότερο βαθμό πολιτική ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών εταιρική σχέση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Από την άλλη, τι ε, κρατά σε επίπεδο προενταξιό. Η εταιρική σχέση υπό την παρούσα μορφή ε, θεωρείται με αυτόν τον τρόπο ότι είναι μια κάποια εναλλακτική αντί να είναι πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 10 χρόνια θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση διότι η διατήρηση της παρούσης καταστάσεως και του παρόντος μοντέλου δεν θα μας οδηγήσει σε επιτυχία. Νομίζω ότι οι ανατολικοί μας εταίροι θα πρέπει να λάβουν ένα σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει να ποντάρουν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Σόκολα, έχετε το λόγο. γιορτάζουμε την επέτειο των 10 ετών για την ανατολική εταιρική σχέση και μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε επιτυχής. Αυτό το τμήμα της Ευρώπης είναι ένα κομμάτι όπου συγκλίνουν τα συμφέροντα των υπερδυνάμεων και εκεί έχουμε 75% της ενέργειας των ενεργειακών πόρων. Μεγάλοι παίκτες έχουν συμφέροντα εκεί και προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθορίσει τα συμφέροντά της στην περιοχή. Έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναστροφή που έχει ξεκινήσει, μια οπισθοχώρηση, μια διολίστηση προς τα, προς τα κάτω όσον αφορά τα δημοκρατικά επιτεύγματα και τα πράγματα δεν είναι όπως θα τα επιθυμούσαμε. Λοιπόν, τρία μηνύματα θα ήθελα να αποστείλω σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε στην ανατολική, ανατολική εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλά με μια φωνή, αυτό πρώτα απ' όλα. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε ατομικά συμφέροντα ή μεμονωμένα συμφέροντα κρατών μελών ε, να αποσυντονίζουν την όλη προσπάθεια, να αποτελούν παραφωνία. Πρέπει να καθορίζουμε κοινά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σαν παγκόσμιο ηγέτη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, πρέπει να δηλώσουμε σαφώ ποια είναι τα συμφέροντά μα, να είμαστε διαφανεί γι' αυτό και να συνομιλούμε με τι φιλοευρωπαϊκέ δυνάμει στι διάφορε αυτέ χώρε. Και τρίτον, ε, θα πρέπει να τηρούμε το λόγο μας. Αυτά που υποσχεθήκαμε. Θα πρέπει να αμείβουμε τα επιτεύγματα που κάνουν αυτές οι χώρες και θα πρέπει να τους δείξουμε ποιος είναι ο καθαρός δρόμος προς την ένταξη. Πρέπει λοιπόν να ανταμείψουμε τις προσπάθειές τους. Ό,τι θεωρούμε ότι είναι φιλοευρωπαϊκό, επίσης τα, την επίτευξη διαφόρων προδιαγραφών όσον αφορά το κράτο δικαίου, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλε άλλε τι μορφέ ελευθερία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για σοσιαλιστικούς δημοκράτες. Η κυρία Μπένοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη για το έργο που έχετε επιτελέσει τη τελευταία πενταετία για όλες αυτές τις προσπάθειες και τώρα θα ήθελα να μιλήσω στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Παρακαλώ να δείξετε ευθύνη στο μέλλον δεν μπορούμε, δεν έχουμε περιθώριο να μην είμαστε θετικοί προς τους ε, γειτόνους μας. Ε, η διαδικασία προσχώρησης της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας σταμάτησαν. Δεν είναι καλή ιδέα αυτή, ειδικότερα στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας. Ε, είναι αποθαρρυντικό για αυτούς ε, αποθαρρυντικό και για τους υπόλοιπους ε, ανατολικούς μας εταίρους. Χρειαζόμαστε μια σταθερή εταιρική σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τη σταθερότητα, την ευημερία, την ασφάλεια. Η συνεργασία με τους ανατολικούς μας εταίρους είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, ιδέες, απόψεις οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης ε, και αυτή η συμφωνία εταιρική σχέση προωθεί τι αξίε που θέλουμε εμεί να υπερασπίσουμε στον κόσμο. Αυτέ οι χώρε ε, κοιτούν με θαυμασμό την ε, Ευρώπη. Οπότε δεν πρέπει να δράμε αρνητικά προ αυτέ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Ντούδα, εκ μέρου του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο των χωρών της Ανατολικής Γειτενίας παρά τις κάποιες δυσκολίες που αναφέραμε εδώ ειδικότερα στη Γεωργία, στην Ουκρανία και στη Μολδαβία καθώς προχωρούν στον δρόμο για την ευρωπαϊκή ε, ένταξη και η Ευρώπη θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι εκτιμά τις προσπάθειές τους. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω τη στρατηγική του τρίου ε, προεδριών για μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικές, ε, επενδυτική στήριξη. Δεν είναι κάτι εύκολο και οι μεταρρυθμίσεις επίσης δεν είναι κάτι εύκολο, το γνωρίζουμε και εμείς. Γι' αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ανατολικούς μας γείτονες. Και ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ στην Ουκρανία, θα ήθελα να συγχαρώ τις νέες αρχές για το θάρρος που έχουν δείξει, διότι οι αλλαγές ε, που εφαρμόζουν ε, ήταν πολύ αναμενόμενες από τους ευρωπαϊκούς εταίρους και από την κοινωνία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, η υπεύθυνη διακυβέρνηση, όλα αυτά είναι μεγάλες προκλήσεις. Η αποκέντρωση και η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών είναι κλειδιά για την ανάπτυξη της Ουκρανικής Δημοκρατίας. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν ευρείες διαβουλεύσεις όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και όλες οι σχετικές οργανώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κοινωνική αποδοχή και για την αποτελεσματική υλοποίηση, αλλά και για την ε, βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ θετικό που η Ουκρανία συμμετέχει σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+. Εγώ έχω συναντηθεί με καταπληκτικούς φιλόδοξους ε, Ουκρανούς νέους και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο χάρη σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συναδελφός Πόσπισιλ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ ήθελα να πω ότι είμαι ικανοποιημένο που μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η εταιρική σχέση. Ενθυμούμε τις συζητήσεις οι οποίες είχαν γίνει πριν από αρκετά χρόνια. Τότε ήμουν μέλος της κυβέρνησης της Τσεχίας και είχαμε προσπαθήσει να παίξουμε κάποιο ρόλο παρόλη την πίεση την οποία εκείνη την εποχή μας ασκούσε η Ρωσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες γειτονίας, ανατολικής γειτονίας, διότι τότε δυστυχώς η Ρωσία, η οποία είναι ήδη ισχυρή σε χώρες όπως η Μολδαβία, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, θα έλεγα Έχουμε να κάνουμε με χώρες των οποίων ο λαός θέλει να ζήσει στη δημοκρατία, σε μια χώρα δημοκρατική και επιμερούσα. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τα δημοκρατικά κοινοβούλια. Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, θετική εκτιμάται γενικά η ανατολική γειτονία και πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία. δεν έχουν άλλη δυνατότητα οι χώρες αυτές. Μεταξύ τους άλλωστε έχουν και διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης και το θέμα της διαφορετικής κάθε φορά παρουσίας της Ρωσίας. Γι' αυτό πρέπει να τις βοηθήσουμε και να τις ενισχύσουμε. Ευχαριστώ. Έχουμε eh, την διαδικασία Catch the Eye. Κλείνει ο κατάλογος με τους ήδη εγγεγραμμένους. Ο, ο πρώτος ομιλητής, σοσιαλδημοκράτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιδράσει για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια ε, είχαμε δυσάρεστες όταν αρνήθηκε το Συμβούλιο τη Σύνεξη της Διαδικασίας Προσχώρησης για αυτές τις ε, χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη αυτές τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Δεν μπορεί να τις ε, κινδυνεύει Αλλιώς θα πέσουν στα χέρια Ρωσίας, Ιράν, άλλων χώρων. Γι' αυτό το λόγο εμεί θα έπρεπε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να παγιώσουμε καλύτερα αυτές τις σχέσεις αυτό είναι προς το καλό των δικών μας λαών. Για την πολιτική της Ανατολικής Γειτονίας η λέξη κλειδί είναι η αρσή των διαφορών. Θα πρέπει ε, αλλά να αναγνωρίζουμε και τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Όταν έχουμε σχέσεις σύνδεσης και καλές εμπορικές σχέσεις, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια οι σχέσεις να εμβαθύνονται. Αυτό προς όφελος όλων των μερών για κάθε μία από τις χώρες, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν. Για όλες αυτές τις χώρες θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια θέση στην πολιτική μας και να προωθήσουμε μεταρρυθμίσει όπως το δικαστικό και να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από την ΚΟΕ, ο κύριος Βόλα uh, um, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μοκερίνη, είπατε ότι η Ανατολική Γειτονία δεν είναι εναντίον κανενός. Παραδέχεστε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και η ανάμειξη επίση της Ευρώπης έχουν ένα στοιχείο κατά της Ρωσίας. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το γνωρίσει αυτό. Δεν πιστεύετε ότι εάν παρέμβαινε στον Καναδά στο Μεξικό η Ρωσία θα υπήρχαν επίσης ε, μεγάλες εντάσεις. Δεν πιστεύετε ότι ήρθε ο η Ευρώπη να εργαστεί για την ειρήνη με τη Ρωσία. Ήταν εταίρος μας. Ειρηνική και έχει πολύ περισσότερο νόημα να προσπαθούμε να κάνουμε ειρήνη με τη Ρωσία και να εμπλέξουμε και τις ε, χώρες που βρίσκονται στην περιοχή να γίνουν ανεξάρτητες ώστε να μην χρειάζονται ούτε τη Ρωσία ούτε τη Δύση. Εδώ πέρα ε, μπαίνουμε σε μια άλλη κούρσα εξοπλισμών. Αντίθετα, πρέπει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Δεν συμφωνούμε σε πολλά, να ξέρετε κυρία Μογκερίνη, αλλά θα μου λείψετε. Ευχαριστούμε. Τσίβαντορ, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής καλείται η δική μου χώρα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ανατολικής γειτονίας, μπορεί να βοηθήσει την δημοκρατία της Μολδαβίας στον τομέα της κατάρτισης της επαγγελματικής και με πάρα πολλά διαμεθοριακά προγράμματα, διασύνοριακά προγράμματα και μάλιστα έχουν καταφέρει να έχουν ακριβώς τα ίδια συστήματα τηλεφωνίας κινητής με το ίδιο κόστος της περιαγωγής με την Ρουμανία. Έτσι μπορούμε να εμπνεύσουμε εκ νέου τους κατοίκους των χώρων αυτών και των περιοχών αυτών με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Να τους οδηγήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντας προγράμματα όπως τον μεγάλο λεωφοριόδρομο ανάμεσα στις διάφορες μεγάλες ρωμανικές πόλεις. Τελευταίος που έχει το λόγο η κυρία Βόρντ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Αυτή τη βδομάδα ο Λαξ ήρθε για να παρελάβει το βραβείο του Σαχάρο που το επενημήθη το 2018 Ξέρουμε όμως ότι κάθε μέρα οι Ουκρανοί πληρώνουν μεγάλο τίμημα για να υποστηρίξουν την εδαφική τους ακαιρεότητα. Υπάρχει πόλεμος στην ανατολική μας γειτονία και αναφέρεται συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης. Η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι 13.000 άνθρωποι και περισσότεροι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στον Ντομπάσκ. Η παράνομη πασάρτηση της ε, Κρυμαία είναι ντροπή για όλου εμά που νοιαζόμαστε για τη δημοκρατία και είμαι περήφανη που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ουκρανία και την επιθυμία της να βρεθεί πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το 2011 εγώ συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα πολιτιστικών ανταλλαγών με Ουκρανούς. Αγάπησα τη χώρα και τον ε, λαό, τους Ουκρανούς. Έμαθα πολλά έμαθα για τη γενοκτονία η οποία σκότωσε 7 εκατομμύρια Ουκρανούς. Η Ρωσία συνεχίζει να κακοποιεί την Ουκρανία και υπάρχει μια ομάδα φίλων της Ουκρανίας. Ποτέ δεν ήταν η καταλληλότερη στιγμή για να δείξουμε όλοι ότι νοιαζόμαστε για την Ουκρανία. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μογκερίνη. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή πιστεύω δείχνει άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι το κοινοβουλευτικό έργο στο πλαίσιο αυτών των εταιρικών μας σχέσεων όχι μόνο με τους ανατολικούς μας εταίρους αλλά και με τους λοιπούς που έχουμε ανά τον κόσμο. Εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο παίζει ρόλο κλειδί όσον αφορά συγκεκριμένα την ανατολική εταιρική σχέση τόσο οι έξι αυτέ χώρε τη εταιρική σχέση, αλλά και πιο συγκεκριμένα το κοινοβουλευτικό έργο που έχετε ε, επιτελέσει εσεί και το έργο που έχετε κάνει με την κοινωνία των πολιτών και του κοινωνικού εταίρους αυτών των έξι συγκεκριμένων χωρών ε, έχει ως αποτέλεσμα τεράστια προστιθέμενη αξία. Και το μόνο που έχω να πω φυσικά είναι λίγο ασυνήθιστο να το συζητάμε τώρα εδώ γιατί φυσικά πλέον δεν μπορώ να σας δεσμευτώ για τα μελλοντικά βήματα θα αφήσω αυτό το καθήκον στα σοφά χέρια του διαδόχου μου της επόμενης επιτροπής αλλά είμαι βέβαιο ότι η οδός που έχει δενεχθεί ε, και που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια ε, για την εμβάθυνση της εταιρική μας σχέσης σε όλους τους τομείς ε, με τις έξι χώρες της ανατολικής εταιρική σχέσης θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον και είμαι βέβαιη ότι θα έχει την πλήρη σας υποστήριξη. Όπως είχα και εγώ την τιμή να έχω τη δική σας υποστήριξη στο έργο μου. Με τις συμβουλές σας, με τις προσπάθειές σας, το έργο σας. Πολλοί από εσάς με ευχαριστήσατε για αυτή την εταιρική σχέση. Θα ήθελα να σας το ανταποδώσω και εγώ ευχαριστώντας εσάς. Διότι πιστεύω ότι δείξαμε ότι πράγματι παρότι μερικές φορές διαφωνούμε από άποψη προοπτικής, αλλά ξέρετε αυτό είναι το θετικό της δημοκρατίας. Μπορείς να διαφωνείς σε κάποια σημεία, παρόλα αυτά συνεχίζεις να κινείσαι προς την ίδια κατεύθυνση σε κάποια άλλα ζητήματα και πιστεύω ότι ιδιαίτερα στην Ανατολική Εταιρική Σχέση αποδείξαμε ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να εργαστούν ενωμένα και να γεφυρώσουν τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Φυσικά ευχαριστώ πολύ για αυτά τα πέντε χρόνια, για την υποστήριξή σας όλο αυτόν τον καιρό και θα παραμείνουμε σε επαφή φυσικά όπως ανέφερα στην προηγούμενο πρόεδρο. Θα παραμείνω μαζί σα το υπόλοιπο βράδυ και αύριο. Οπότε α μην αποχαιρετιστούμε ακόμα. Δεν είναι τα τελευταία λόγια αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εδώ κλείνει λοιπόν η συζήτηση για τις εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι μια δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή ΥΠΑ τη Εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία για την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά του οικισμού. Έχετε και πάλι το λόγο, κύριε Μουγκερίνη. Uh, Ξεκινώντας, θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι μαζί. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά αυτή εδώ και πέντε χρόνια και λίγες εβδομάδες, η πρώτη μου επίσκεψη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, επισκέφθηκα και τη Λωρίδα της Γάζα και είπα ότι τότε θα μπορούσαμε να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της εντολής μου τη λύση των δύο κρατών. Αυτός ήταν ο στόχος ο οποίος με ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά την οποία έκανα Μερικές φορές ο στόχος αυτός φάνηκε να είναι εγκύτερος, αλλά δυστυχώς η κατάσταση σήμερα είναι το αντίθετο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον η προοπτική αυτή. Είναι θέμα, θα έλεγα, πολιτικής βούλησης, αλλά σήμερα αυτό το οποίο είναι σαφές, ότι δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξοι Η ιδέα των δύο κρατών είναι κάτι το οποίο είναι στο νου πάρα πολλών και ακόμα και εμπλεκομένων σε αυτή τη διαφορά. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε κάποιες ρεαλιστικές λύσεις. Θα έλεγα ότι η λύση των δύο κρατών είναι μια ρεαλιστική λύση κανένας δεν έχει προτείνει ε, στην λύση αυτή μια εναλλακτική αξιόπιστη. Πολλοί κατακρίνουν την λύση των δύο κρατών. Κανείς όμως δεν είναι σε θέση ρεαλιστικά να εκφράσει, ε, θα έλεγα, μια εναλλακτική λύση και σε επίπεδο διεθνού συνταγματικού δικαίου και σε επίπεδο πεπιθήσεων και των κατοίκων της περιοχής ε, δεν υπάρχει μια άλλη λύση. Το θέμα λοιπόν είναι και διεθνώς, διεθνούς δικαίου θέμα, είναι θέμα δημοκρατίας και είναι όπως είπα και θέμα πραγματισμού. Έκανα κάθε προσπάθεια ε, τα τελευταία χρόνια για να διατηρήσω την προοπτική των δύο κρατών, της λύσης των δύο κρατών και συνεχίζω και σήμερα κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ε, όπως βλέπω ότι πολλοί φίλοι στην περιοχή και κάποιοι ακόμα μακρύτερα ε, οι φωνές του ρεαλισμού και ε, της σοφίας δεν ακούγονται τόσο δυνατά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο αντικειμενικός στόχος δυστυχώς απομακρύνεται. Αυτό πρέπει να μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο επίμονοι και ακόμα ταχύτεροι. Αυτές είναι οι θέσεις μας και για το θέμα των επικισμών. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αλλαγές στα σύνορα μπορεί να αποφασιστούν με άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη με βάση τα σύνορα που είχαν αποφασιστεί παλαιότερα. Οι εγκαταστάσεις αυτές του Ισραήλ είναι παράνομες σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και δυστυχώς καθιστούν αδύνατη την προοπτική της λύσης. Επίσης οι θέση του Ισραήλ για την Ιερουσαλήμ ε, δημιουργεί προβλήματα στην λύση της Ιερουσαλήμ πόλης πρωτεύουσας και για τις δύο χώρες. Συνεπώς λοιπόν ε, θυμίζω ότι πάντα είχαμε μια ενωμένη ευρωπαϊκή θέση. Σε δύσκολες στιγμές η Ευρώπη στο συγκεκριμένο θέμα έχει μια ξεκάθαρη ισχυρή και ενιαία θέση. Και φυσικά εδώ δεν αγνοούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. Οι ε, επιθέσεις με πυράβλους μικρού πελληνικού εις του Ισραήλ είναι απαράδεκτες και τις καταδικάζουμε. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην ασφάλεια. Οι πολίτες του Ισραήλ έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ασφάλεια θα είναι βιώσιμη και πραγματική όταν αδράζεται ακριβώς την λύση των δύο κρατών. Προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια επίσης να ελαφρύνουμε τα βασανιστήρια τα, οποία υποφέρει ο λαός της Γάζα και σε επίπεδο σχολείων, νοσοκομείων, υποδομών. Η κατάσταση στην Γάζα είναι προβληματική και σε επίπεδο πολιτικό. Πρέπει ο αποκλισμός να τελειώσει πλέον και να ανοίξουν οι δίωδοι. Είναι σαφές επίσης ότι η Γάζα ανήκει στο νέο ε, Παλαιστινιανό κράτος στα πλαίσια της λύσης των δύο κρατών και οι Παλαιστίνοι πρέπει συνεπώς να ξεπεράσουν τις διαιρέσεις τους. Θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι επαφές ανάμεσα στα δύο μέρη. <clears throat> Η Παλαιστινιακή πλευρά ανακοίνωσε ο Αμπάς εκλογές πρόσφατα η Ισραηλινή πλευρά βρίσκεται σε αδιέξοδο σε επίπεδο κυβερνητικό και μπορεί να γίνουν ξανά εκλογές για πολλωστή φορά μέσα σε ένα χρόνο. Επιμένω, η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις είναι πιθανή πέντε χρόνια μετά την πρώτη μου επίσκεψη πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και μπορούμε να το πετύχουμε γιατί είναι η μοναδική βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για το Μεσανατολικό. Είμαι επίσης προσωπικά πεπισμένη ότι από όλε τις συγκρούσεις της περιοχής ή το πρόβλημα αυτό είναι το πιο εύκολο που μπορούμε να λύσουμε εφόσον βέβαια υπάρχει αυτό που είπα στην αρχή, η πολιτική βούληση ανάμεσα στις χώρες και ανάμεσα στους διεθνείς εταίρους. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη αν δεν υπάρχει πραγματική προσπάθεια και αφοσίωση για λύση. Εμείς στην Ευρώπη πάντα και εξακολουθούμε και σήμερα να στηρίζουμε και να συνοδεύουμε κάθε μέτρο που στοχεύει στην ειρήνη και στην διαπραγμάτευση για τη λύση των δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μογκερίνη. Τώρα, οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα, πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Λόπες Αστούριθ Βάιτ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, ε, κυρία Αντιπρόεδρε. Θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να σας ευχαριστήσω για αυτά τα πέντε χρόνια ε, πραγματικών ανταλλαγών ε, απόψεων μεταξύ μας. Και τώρα για το θέμα της Παλαιστίνης είμαι σίγουρος ότι είναι από τα πιο δύσκολα θέματα που είχατε να χειριστείτε κατά τη θητεία σας. Και να ξέρετε ότι σας στηρίζουμε και συμμερίζομαι ε, πολλά από αυτά τα οποία είπατε. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν πρόκειται να λυθεί γρήγορα, αλλά όλοι καλή τη πίστη συμμετέχουμε και προσπαθούμε από κάθε πλευρά να υπάρξει μια λύση και μια σταθερότητα, όχι μόνο για αυτή τη σύγκρουση που ταλαιπωρεί αυτή την περιοχή, αλλά και γενικότερα ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας. Τώρα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να πω ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα στρατηγική σημασία σε τέρο μας και έχουμε κοινή ιστορία και κοινέ αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ είναι δημοκρατίες και προσπαθούμε τις δικές μας τις αρχές και τις αξίες να τις προωθήσουμε ανά το κόσμο υπέρ του κράτους δικαίου για άλλες χώρες και λαούς. Υπάρχει ανησυχία στο Ισραήλ για την ασφάλειά του και είναι λογικό. Είδαμε ε, τις εκτοξεύσεις που έγιναν πρόσφατα και καλό είναι να μην υπάρχει κλιμάκωση και χαιρετίζουμε ότι αν μη τι άλλο σταμάτησαν αυτέ οι επιθέσεις. Εμείς πάντω δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο σε δηλώσει, γιατί πάντα έχω την αίσθηση ότι μιλάμε και ακολουθούμε τους Αμερικανούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν αντιδρά από μόνη τη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς στο διάλογο και στην ειρήνη με τον δικό μας τρόπο δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε από τα διάφορα tweets και τις διάφορες δηλώσεις. Είναι σημαντικό να εργαστούμε, να έρθουν ε, βουλευτές ε, βεβαίως από την Κνεσέτ και θα έρθουν νομίζω σε μερικές εβδομάδες εδώ στο Στρασβούργο αλλά και σε εκτελεστικό επίπεδο οι υπουργικέ ε, συναντήσεις που διακόπησαν να συνεχιστούν και να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Έπειτα, το έργο μας όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων που μας έρχονται από τους επικισμούς είναι ένα σφάλμα. Αντίθετα, θα έπρεπε να συνεργάζεται με το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η ανάπτυξη στην περιοχή. Θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα προσέγγιση που να προσφέρει μεγαλύτερη ευημερία στην περιοχή. Έτσι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε να τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Τώρα για κάποιους κομμουνιστές ε, που γελάνε. Ωραία, θα σας ακούσω, αλλά εγώ δεν θέλω εδώ πέρα να προσβάλλω κανέναν, δεν τα βάζω με κανέναν. Απλώς πιστεύω ότι μπορούμε απέναντι στους Ιρλανούς και τους Παλαιστινίου να βοηθήσουμε να υπάρξει εκεί προσέγγιση. Και θα το είδατε, σε αυτά που είπα δεν επιτέθηκα ε, στην ε, Παλαιστίνη για να ακούσουμε τι θα πούνε και άλλοι και αν θα επιτεθούν. Ευχαριστώ. πολύ. Η κυρία Πύρη έχει το λόγο. Ε, κυρία Επέτη, εκπρόσωπα, αγαπητοί συνάδελφοι, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις πρόσφατες δηλώσεις των ΗΠΑ μετά από το γύρο συγκρούσεων, βίων συγκρούσεων, ο Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο ανακοίνωσε αλλαγή τη Αμερικανική πολιτική όσον αφορά του Ισραηλινού επικισμού. Είπε ότι η εγκατάσταση ε, μη στρατητικών οικισμών του Ισραήλ στην Λωρίδα Γάζα, δεν, στην περιοχή αυτή, δεν ε, είναι παράνομη, παρότι παραβιάζει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, και την απόφαση του Διεθνούς ε, ε, Δικαστηρίου. Υποστηρίζω να έχετε μία αντίδραση άμεση, κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε. Η Ισραηλινή επικισμοί είναι παράνομη υπό το Διεθνές Δίκαιο και το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να τερματίσει όλε τι διαδικασίε επικισμού και δραστηριότητε επικισμού ω δυναμή κατοχή. Η ανακοίνωση του Πομπέου είναι άλλη μία Άλλο ένα παράδειγμα της αιμονής ε, υπέρ του Νιατανιάχου από πλευράς του Τραμπ ε, ακολουθεί την ανακοίνωση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα στην ε, μεταφορά της Αμερικανικής πρεσβείας και την αναγνώριση των υψηπέδων του Κολάν. με την συμφωνία του αιώνα όπως την ονόμασε ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να κλιμακώσει τη σύγκρουση ει βάρο των Παλαιστινίων, των Ισραηλινών και τη ε, διεθνού κοινότητα. Ο πρόεδρο Τραμπ πρέπει να καταλάβει ότι η Μέση Ανατολή δεν είναι ε, χώρο όπου αυτό μπορεί να ασκεί την εξωτερική του πολιτική. Είναι σπίτι για εκατομμύρια ε, παλαιστινίου και Ισραηλινούς που παλεύουν για την ειρήνη καθημερινά. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στην Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σαφώ υπονομεύει την προοπτική οποιασδήποτε βιώσιμη λύση δύο κρατών η οποία είναι η μόνη ελπίδα για βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Υπό αυτό το πνεύμα υποστηρίζουμε και την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την επισήμανση των προϊόντων από ε, περιοχές επικισμών στις αγορές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βάλτμαν. Η κυρία Βάλτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, Πρώτα απ' όλα θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια που ήρθατε εδώ τόσο συχνά και ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ καθόσαστε και συζητούσατε μαζί μας. Τώρα συζητάμε για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, όπως τόσες και τόσες φορές μέχρι σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη στην τελευταία θητεία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ξανά και ξανά. Γιατί το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει 12.000 κατοικίε στην Παλαιστίνη και από το 2009 6.000 κτίρια στη Δυτική Όχθη έχουν καταστραφεί. Και μάλιστα που έχουν χρηματοδοτηθεί και χτιστεί με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Το Ισραήλ βήμα-βήμα προχωράει για να δημιουργήσει μια πραγματικότητα του ενός κράτους. Και δεν θα υπάρχει πια περιθώριο κανένα για τους Παλαιστινίους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Η Ευρώπη λέει ότι είναι υπέρ του κράτους δικαίου, ότι βασίζεται στο δίκαιο. Οπότε και εμείς πρέπει να τα βάλουμε με την πολιτική δύναμη του Νετανιάου, να τα βάλουμε με την πολιτική επικισμών. Εμείς, η Ευρώπη, πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη λύση αυτή των δύο κρατών, που για μένα είναι η μόνη λύση. Η... Κύριε, είπατε εκπρόσωποι, φαντάζομαι ότι είναι τελευταία σα, η μία από τι τελευταίε παρεμβάσει σα εδώ στο Στρασβούργο. Αλλά είπατε ότι θα παρακολουθείτε τι γίνεται και τι ε, λύσει που θα βρεθούν στο μέλλον. Πρέπει Κάθε φορά που καταστρέφονται δικά μας προγράμματα πρέπει να αντιδράμε, όπως είπατε και εσείς, και να ε, υψώνουμε τον αίσθημά μας κατά του Τραμπ ή του Νιαταγάου όταν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Ε, κυρία, είπατε εκπρόσωπε, αν το κάνετε αυτό, έχετε και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην μελλοντική σας σταδιοδρομία ή οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ο μιλητή, ο κύριο Σάλιβαν, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε, κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε. Η κίνηση τη δίκηση Τραμπ για την αναγνώριση των παρανόμων επικισμών στη Δυτική Όχθη είναι το τελευταίο επεισόδιο στι πολύ ανησυχητικέ παρεμβάσει μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει να καταστρέψει οποιαδήποτε ευκαιρία ευκαιρία ε, ειρήνη ε, Αναγνωρίζοντας τις παράνομες, ε, τους παράνομους επικισμούς, ε, οι ΗΠΑ παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζουν εκείνους που προσπαθούν να διασφαλίσουν ε, μη βιώσιμο μέλλον μεταξύ των δύο κρατών. Είναι αδιαμφισβήτητη η παρανομία. Οποιαδήποτε χώρα προσπαθεί να επικίσει εδάφη που έχουν αποκτηθεί μέσω συγκρούσεων πραγματοποιεί παρανομία. Πιστεύω ότι όλοι επιθυμούμε να υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση που θα εκπροσωπεί και θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Κάθε βήμα κατοχής προσάρτησης είναι ένα βήμα που μας απομακρύνει από μια διπλή σταθερή κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον. Γνωρίζουμε ότι η ΕΠΑ δεν είναι και δεν πρόκειται να είναι αξιόπιστος εταίρος στη διαδικασία αυτή διότι όσο η τρέχουσα διοίκηση διοικεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει μια βιώσιμη λύση για την περιοχή και που μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ειλικρινής για την ειρήνη. Δεύτερον, πρέπει να δούμε πώς εμείς ως Οικονομική Ένωση θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Δεν θέλω και δεν πρόκειται να ε, υποστηρίξω ε, το κίνημα επιδίας, αλλά ούτε ε, τις δραστηριότητες σε κλεμμένη γη που έχει προσαρτηθεί με παραβίαση του διεθνούς δικαίου ο γερουσιαστής Μπλακ ε, ε, ε, σε εμά στην Ιρλανδία αποφάσισε να απαγορεύσει προϊόντα που παράγονται σε αυτές τις επικισμένες περιοχές και εγώ το υποστηρίζω. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μα όπου έχει ληφθεί βάση τη Σύμβαση τη Γενέβη. Τα προϊόντα που παράγονται στι παράνομε επικισμένε περιοχέ στη Δυτική Όχθη εισάγονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο, μέρος, στο πλαίσιο μια εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ που δεν εκτείνεται και σε αυτέ τι περιοχέ Θέλω να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να επιτρέπετε να συνεχίζετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φέστ, έχετε το λόγο εκ μέρου του κόμματο Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, λέτε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη, η πιο βιώσιμη, η πιο ρεαλιστική. Το αντίθετο όμως ισχύει η λύση των δύο κρατών δεν είναι μια έκφραση της πολιτικής άγνοιας και της απώλειας του ρεαλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο κράτη σημαίνει να δοθεί η Δυτική Όχθη και η Γάζα πίσω σε αυτούς και αυτό θα φέρει ειρήνη. Όχι. Το 2000 ήδη ο Γιάσερ Αραφάτ είχε κάνει μια γενναιόδορη, είχε αρνηθεί μια γενναιόδορη προσφαρά. Ο Μαχμουνταμπάς έκανε το ίδιο αργότερα και το Ισραήλ το 2005 ε, υποχώρησε και παρότρινε τη Χαμάσα να ελευθερώσουν τελείως την ε, Παλαιστίνη. Ε, η Χαμάς και η Αλφατάχα δεν πρέπει να βρίσκονται ούτε στη δική ούτε στην ε, Γάζα. Βρίσκονται και στη Χάιφα και παντού. Και στην Ιερουσαλήμ τελικά. Κυρία Μογκερίνη, μιλήσατε για πολιτική βούληση η οποία απαιτείται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ, επιτέλους, αντιληφθείτε από πλευράς των Παλαιστινίων της Παλαιστινιακής Αρχής. Αυτή η βούληση δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει και γι' αυτό τον λόγο η δική σας πολιτική των δύο κρατών της λύση αυτής είναι λανθασμένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος είναι ο κ. Ράισεν από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατή εκπρόσωπε. Δήλωση του κυρίου Πεμπέου ε, δημιούργησε βέβαια πολύ φασαρία. Στο μεταξύ όμως έχουν κάποιο δίκιο, γιατί το να λέμε ότι είναι παράνομοι επικισμοί είναι μεγάλα λόγια. Δεν μπορούμε να ανταμείβουμε τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ ιστορικά αλλά και νομικά έχει το δικαίωμα να χτίζει στην περιοχή. Οι επικισμοί και ο χώρος στον οποίο χτίζονται είναι χώρος που αμφισβητείται για το σε ποιον τελικά νίκη. Οπότε συμφωνώ ότι πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει να επενδύουμε αντί να τσακωνόμαστε. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Γιατί έτσι θα βοηθήσουμε την περιοχή και έτσι θα τη φέρουμε και πιο κοντά μας. Γι' αυτό και λέω να σταματήσουμε να στηρίζουμε τους τρομοκράτες και τις οικογένειες τους μέσω της Παλαιστινιακής κυβέρνησης, όπως κάνει η Ολλανδία. Να σταματήσουμε να πληρώνουμε την Ούνρα, η οποία έχει οδηγήσει σε μια φοβερή κατάσταση. Και να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά το Ιράν, που έχει επιθετική συμπεριφορά στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πινέντα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να συγχαρώ την κυρία Μογκερίνη για αυτά που είπε μετά τις δηλώσεις Πομπέο που μίλησε για τους παράνομους επικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Και θέλω να τη συγχαρώ για το περιεχόμενο της δήλωσής της, αλλά και για το ότι την έκανε αμέσως. Και θέλω να σημειώσω ότι πάντα το έκανε αυτό κατά τη διάρκεια της εντολής της. Ελπίζω και είμαι πεπισμένος ότι το ίδιο θα κάνει και ο κύριος Μπορέλ. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε κυρία Μογκερίνη για το ότι παρόλο που η δήλωση και όλε οι δηλώσεις που κάνατε ήταν πάντα καλές και είχαν αξία γιατί βέβαια ε, δείχνουν ότι δεν συμφωνούμε με τις συνεχείς παραβιάσεις του Ισραήλ παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι δεν είχε και μεγάλο εφέ. Γιατί το θέμα είναι ότι είναι γενναιόδοροι οι Παλαιστίνοι και προσφέρουν 68% της επικράτειάς τους και ε, δέχονται ότι είναι κράτος, ενώ στο υπόλοιπο 22% δεν μπορεί να υπάρξει κράτος. Μα είναι δυνατόν. Το Ισραήλ συμφωνεί με το με το, το λέει ο ΙΕ. Τώρα, τι παράδειγμα μπορώ να πω για το Ισραήλ, ότι συστηματικά παραβιάζει. Και η τελευταία επίθεση, ο Νετανιάου πώς λύνει τα προβλήματα με βομβαρδισμούς. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, λέει ο Πρόεδρος. Ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ, δώστε μου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να την αναγνωρίσει ως κράτος και να πιέσουμε και τις χώρες μέλη να κάνουν το ίδιο. Και να σταματήσουν οι συμφωνίες, διακόπτη Πρόεδρος. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να τηρούν το χρόνο τους, παρακαλώ σεβαστείτε τους συναδέρφους σας και μην ξεπερνάτε το χρόνο σας, παρακαλώ. Επόμενος ο μιλητής, Φόρμαν. μία εγγεγραμμένος. Είναι ψέμα να λέμε ότι είναι παράνομοι οι επικισμοί Ισραηλινοί, αμφισβητούμενοι, αλλά παράνομοι δεν είναι ήδη από τις παλαιές συμφωνίες, ήδη από τη συμφωνία του 1922 ε, δεν ε, έχει υπάρξει κάτι παλαιότερο και έτσι και αλλιώς και η Δυτική Όχθη είναι τμήμα του Ισραήλ. Ποτέ δεν ήταν ανεξάρτητη χώρα. Όταν έφυγαν οι Βρετανοί το 1948 ξέσπασε πόλεμος και ε, φυσικά η όχθη αυτή κατακτήθηκε από την Ιορδανία αλλά η εισβολή αυτή δεν φυσικά έγινε δεκτή από κανένα. Οπότε το 67 το Ισραήλ ανακτώντας το έδαφος δεν διέσχισε διεθνή σύνορα. Στην ουσία λοιπόν παρεμεινεύεται το 49 τη σύμβαση της Γενέβης. Εδώ και δύο εβδομάδες ε, υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να βάζει διαφορετικές ετικέτες ε, στα προ... υποχρέωσε το Ισραήλ και τους επίκους διαφορετικές ετικέτες από ότι η παραγωγή το υπόλοιπο Ισραήλ. Αυτό είναι παράλογο ε, γιατί δεν είναι νομικά αποδεδειγμένο ότι είναι παράνομη η συγκεκριμένοι οικισμοί. Η λογική είναι ότι λέγοντας συνεχώς ψέματα κάποιος θα σε πιστέψει. Καιρό είναι να αλλάξει αυτή η λογική και τότε μόνο με την αλήθεια θα πετύχουμε την ειρήνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Σόφκο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. για αυτά που είπατε για την ειρήνη ε, στη Μέση Ανατολή και ανάμεσα στους Παλαιστινίους και το Ισραήλ.